θα πρέπει να σταματήσουμε λίγο νωρίτερα λόγω εκτάκτων περιστάσεων, αλλά πιστεύω πως θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε όλες τις ε, πληροφορίες, να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας που είναι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρία. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στους φακέλους, αλλά σας ε, πω κάποια πράγματα καθώς ε, θα προχωράμε. Καταρχά θέλω να ξεκινήσω ε, κρίνοντας το σχέδιο μερικής διάταξης. Η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Μας ακούτε παρακαλώ στην ελληνική καμπίνα. Ένα μικρό νεύμα. Αν μας, Μα, ακούτε, αν μας ακούτε μπορείτε να μας κάνετε ένα μικρό νεύμα στην ελληνική καμπίνα αριθμός 7. And we will consider them adopted. Um,